αλλά μαζί θα τα καταφέρουμε σίγουρα καλύτερα. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Commissioner. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Μια τελευταία αναγγελία. Η συνεδρίαση διακόπτεται για αύριο 15 Ιουνίου στις 9 μέχρι τις 1 και από 3 μέχρι τις 8.30 και από 9 μέχρι 12 το βράδυ έχει δημοσιευτεί η μέση διάταξη και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ τους Γερμανείς και το προσωπικό. Ολοκληρώνεται η συνεδρίαση.